Σχέδιο σύστασης για την απόφαση του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003-16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το προσαρτημένο πρωτόκολλο στη συνθήκη της ΕΚΑΧ μετά από την λήξη της ισχύω της συνθήκης αυτής και του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλιβα. Είμαι εισηγητής. Θα σας εκθέσω την πρότασή μου. Όταν δημιουργήθηκε το Ταμείο, πήρε τα ενεργά στοιχεία της ε, ΕΚΑΧ περίπου 2 δις ευρώ. Μετά από σοφές θα έλεγα μεταφορές, ε, κάθε χρόνο υπήρχε ένα έσοδο 40 εκατομμυρίων και με τα 47 εκατομμύρια χρηματοδοτούσαμε την έρευνα 72,40% για το χάλιβα και ένα αντίστοιχο ποσοστό για τον άνθρακα. 27,2% για τον άνθρακα αλλά μετά από τις αλλαγές που έγιναν δυστυχώς έπεσε το έσοδο αυτό και τώρα δεν ξεπερνάνε τα 26-27 εκατομμύρια και όχι 40 που ήταν κάποτε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Έχω προτείνει εγώ να χρησιμοποιήσουμε τις υποχρεώσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν, τα αποθεματικά κατά κάποιο τρόπο, για να φτάσουμε στα 40 εκατομμύρια εκ και να αντισταθμίσουμε την μείωση των εσόδων από τόκους μετά την τοποθέτηση σε λογαριασμούς απόδοσης των 2 δις. Πήρα διάφορες γνώμες και συμβουλές από ειδικού. Ε, που ασχολούνται με θέματα έρευνας για ειδικά κράματα χάλιβα και για τον Χάλιβα διάφοροι σύμβουλοι. Ε, είναι περίεργο που κάνουμε έρευνα για τον άνθρακα, αλλά είναι σημαντικό να μειώσουμε την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα με τη χρήση του υλικού αυτού. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ συμφωνώ, πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την πρόταση η οποία γίνεται. Ε, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω θα ήθελα αν έχετε αντιδράσεις να μου τις μεταφέρετε. Ποιος θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ως σκιώδης για την ΚΟΕ Σε τεχνικό επίπεδο και σε σχέση με το δημοσιονομικό θέμα θα συμφωνήσουμε έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το τμήμα αυτό για τα υπόλοιπα της ΕΚΑΧ. Η λύση την οποία προτείνει ο εισηγητής είναι βιώσιμη, αλλά θα πρέπει να εκφράσουμε κάποιες ε, πολιτικές επιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση των ποσών αυτών. Θα θέλαμε να πούμε ότι μιλάμε για δύο τομείς, τον άνθρακα και τον Χάλιβα που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παρούσα φάση για διαφορετικούς λόγους. Ιδιαίτερα για τον άνθρακα είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο διεθνές η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε διαδικασίες ε, για εγκατάλειψη της χρήσης του άνθρακα και έχουν γίνει αρκετά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και γι' αυτό εμείς δεν θεωρούμε ότι οι τεχνολογίες ε, οι οποίες επιδοτούνται μέσω του ταμείου αυτού για, την, ε, για το καθαρό άνθρακα όπως λέγεται ή για, την, ε, για τον περιορισμό των εκπομπών είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβατά με την πολιτική την οποία ακολουθούμε στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι στρεβλές λύσεις προτάσεις για την επίλυση των κλιματολογικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα η βιομηχανία του άνθρακα η οποία δεν περνάει μια καλή φάση στην παρούσα φάση, μια, ε, στην παρούσα περίοδο Πράγματι θα πρέπει να υπάρξει αναζήτηση νέων τρόπων, εκ νέου χρήσης, η ανακύκλωση των υλικών και έτσι να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και ε, να ενισχυθεί η κυκλική οικονομία και στον τομέα του χάλιβα. Λοιπόν, η πρόταση είναι βιώσιμη, αλλά σε πολιτικό επίπεδο έχουμε επιφυλάξεις. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι εμπειρογνώμονες και οι διαχειριστές του ταμείου αυτού θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις παρατηρήσεις σας. Αλλά ταυτόχρονα σημειώνω τη συμφωνία σας με το γενικό προσανατολισμό. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Να πω ότι αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 12 το μεσημέρι την 30 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές και για το σύνολο της έκθεσης θα γίνει στις 21-22 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας και στις 12 Μαρτίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο νομίζω. Η επόμενη έκθεση τώρα. Είναι η, η εφαρμογή των μέσων χρηματοδότησης για την αναθεώρηση και τις αλλαγές μετά το 2020 και έρχομαι εδώ σε αυτά τα οποία είπαμε σήμερα για το επόμενο πολιετές. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας προτείνω είναι να υπογραμμίσουμε ότι το μέγεθος της χρηματοδότησης της κοινοτικής στον τίτλο 4 του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και η έλλειψη ευαισθησίας και ελαστικότητας δείχνει ε, πόσο ε, λίγο φιλόδοξη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει σαν παγκόσμιος εταίρος. Η μείωση γενικά του του Ειδικού Ταμείου για την Τουρκία και ο τρόπος με τον οποίο ε, χρηματοδοτήθηκε μειώνουν την διαφάνεια ε, και μειώνουν και τον ίδιο τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για τις πολιτικές της και νέες πιστώσεις. Η αισθησή μου είναι ότι οι εξωτερικές μορφές χρηματοδότησης μετά το 2020 θα πρέπει να εξυπηρετούν μία και συνολική ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανάλογα με τις φιλόδοξες πολιτικές οι οποίες έχουν αποφασιστεί και επιτρέποντας να υπάρξει μια συνολική πολιτική παρέμβαση της Ένωσης, επιτρέποντας την Ένωση να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη, με υψηλότερη ταχύτητα ε, στις διεθνείς προκλήσεις, να δημιουργηθεί μια προστιθέμενη αξία γιατί η χρηματοδότηση αυτή δεν θα πρέπει να επικαλύπτεται με τα θέματα που προσανατολίζονται στην προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα και να σέβονται, ε, θα έλεγα, τις βασικές αρχές που υπογραμμίσαμε σήμερα το πρωί, δημοσιονομικές αρχές ειλικρίνειας και ενότητας δημοσιονομικής, να αποφύγουμε την παρουσία αυτή του τεράστιου γαλαξία ταμείων που καθιστούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δυσανάγνωστο. Σας προτείνω λοιπόν να απλοποιήσουμε το σύστημα αυτό για να, των εξωτερικών ταμείων για να βελτιωθεί η ορατότητα και η διαφάνεια των ταμείων αυτών και να μπορέσουν και οι βουλευτές και οι ε, φορολογούμενοι να κατανοήσουν το είδος αυτής της αρχιτεκτονικής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα εξωτερικά ταμεία αυτά να ενταχθούν ακόμα περισσότερο στο ε, κεντρικό δημοσιονομικό σώμα της Ένωσης και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσουν ε, περαιτέρω στοιχεία για κάθε αυτόνομη πίστοση. Απαιτείται ευελιξία, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές είναι οι προτάσεις τις οποίες θα ήθελα να σας κάνω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Φερνάντες. Συμφωνώ με τις προτάσεις σας, Πρόεδρε αλλά θα μιλήσω εξ ονόματος του σκιώδους εισηγητού μας για αυτό το θέμα. Τη ο εισηγητριάς μας μάλλον. Και μάλιστα θα μιλήσω πορτογαλικά. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή που μας παρουσίασε τις θέσεις του. Η κυρία Μάλετιτς, η, η σκιώδης σύμφωνη πρόκειται για μια ανάλυση που γίνεται στο ενδιάμεσο, στο μέσο της περίοδου του ε, πολιτικού Διαπιστώνονται, πρόοδος, παρόλο ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα. Η, η, η ε, ζητά να καταγράφονται οι στόχοι κάθε προγράμματος έτσι ώστε να είναι δυνατόν να παρακολουθείτε η αποτελεσματικότητα της διάθεσης των πόρων. Ε, αυτή η αποτελεσματικότητα, αυτή η πρόοδος ε, είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Η συγγήτρια επίση ε, επιμένει στο θέμα της απλοποίησης, όπως είπε και ο εισηγητής. Μετά από το 2020 αυτή η απλοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ενίσχυση των συνεργειών, συνδυασμό της δράσης των ταμείων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Δηλαδή να επιζητούμε πάντοτε μια ε, συμπληρωματικότητα. υπάρχει δυνατότητα να ενσταλλάξουμε και μεγαλύτερη ευελιξία και είναι απαραίτητο για να μπορούμε να αντιδρούμε πιο γρήγορα σε απρόσμενα γεγονότα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης από SND ε, θα ε, ήθελα να συμφωνήσω με αρκετά τα οποία υπόθηκαν, όμως θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα όσον αφορά μεγάλους οργανισμούς όπου υπάρχουν μεγάλοι προϋπολογισμούς, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για ε, διοικητικό χάσιμο χρόνου και θα πρέπει να προσέχουμε σε αυτό. Η έκθεση της Κοπισιόν καταλήγει ότι τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης ε, υπάρχει μια ε, σημεία όπου συμπίπτουν αυτά και, θα πρέπει, και όσον αφορά την ευελιξία την οποία προσφέρουν για τις διάφορες συνθήκες οι οποίες προχύπτουν η συνοχή μεταξύ των ε, μέσων θα βελτιώσει ε, τα όρια μεταξύ θεματικών και γεωγραφικών προγραμμάτων που μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο ε, θέμα όπως ε, για παράδειγμα το Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο συμπίπτει με άλλα θέματα και αυτά είναι σημεία τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί στην έκθεση ευτυχώς ούτε ε, καμία από τις εκθέσεις της ε, Επιτροπής δεν κάνει συστάσεις σχετικά με το πώς αυτές, αυτά τα μέσα και συνεργείες μπορούν να επιτευχθούν στην πράξη, τουλάχιστον για την ώρα. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι ο στόχος ε, τέτοιων εκθέσεων είναι ε, ότι θα χρησιμοποιηθεί όλος αυτός ο χρόνος ε, για να προκύπτουν σχέδια για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις συνεργείες μετά το 2020. χρειάζεται η βελτίωση της ευελιξίας. Ε, θα θέλαμε να αποφύγουμε όμως να επαναχρησιμοποιήσουμε το, ε, τα ποσά για την ανάπτυξη στην ασφάλεια. Πέρσι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε τον προϋπολογισμό ε, χρησιμοποιώντας ε, ποσά 7,2 εκατομμύρια από το μέσο για την ανάπτυξη και τα χρησιμοποίησε αυτά για, για το μηχανισμό για την ασφάλεια. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ικανότητες για να δημιουργήσουμε δημιουργηθούν ικανότητε για την ανάπτυξη. Η ομάδα μα ήταν κατά αυτού και παραμένουμε διότι επαναλαμβάνουμε στι συζητήσει μα ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νέου τομεί όπου εργάζεται, τότε αυτοί οι, τομεί χρειάζονται και νέου πόρου. Και επιπρόσθετα η ανάπτυξη, οποία, ε, θα, ε, τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση τη διαμάχη δεν θα θυσιαστούν για χάρη τη ασφάλεια, αλλά θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τα αίτια που προκαλούν αυτά. Θα πρέπει επίσης να ε, προωθήσουμε τις προτεραιότητες που ευελπιστούμε ότι ε, με, ε, με τους μηχανισμούς για μετά το 2020, 2020 θα επικεντρωθούμε στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να είναι παγκόσμιες αξίες και θα επικεντρωθούμε ιδιαιτέρως σε θέματα τα οποία αφορούν την ισότητα των φύλων στις αναπτυσσόμενες χώρες πρακτικά μέσα όπως για παράδειγμα η σεξουαλική υγεία και η αναπαραγωγική υγεία αυτά είναι δεν είναι πράγματα που είναι ωραία να έχουμε, είναι βασικά ζητήματα ανάπτυξης τα οποία εμποδίζονται από την ε, νομοθεσία του ε, Donald Trump ο οποίος αποτρέπει την ε, αμερικανική χρηματοδότηση τέτοιων ΜΚΟ που υποστηρίζονται τέτοια θέματα. Επίσης, οποιοδήποτε πρόγραμμα το οποίο δεν εκπληρώνει τους στόχους του και τα χρήματα τα οποία δεν δαπανούνται στους σκόπους τους οποίους στοχεύουν θα προτείνουμε λοιπόν ότι, θα πρέπει, ότι υπάρχει χώρος βελτίωσης από ότι ε, αναγνωρίζει η ίδια η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιο άλλο θέλει το λόγο. Κανείς σημειώνει τι παρατηρήσει σα, Κύριε Χάουαρθ. Χρειάζεται πίεση προκειμένου το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο να ενταχθεί στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου η ευρωπαϊκή πολιτική να γίνει πιο ευανάγνωστη, πιο ορατή. Οι τροπολογίε πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τι 2 Φεβρουαρίου, 4 ώρα το απόγευμα. Η ε, ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή θα γίνει στι 21-22 Φεβρουαρίου, ενώ στην ΑΦΕΤ, μια και εμεί μόνο γνωμοδοτούμε, θα γίνει στι 8 Μαρτίου. Περνάμε στην επόμενη έκθεση εφαρμογή του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας, του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, θέμα της ε, Επιτροπής ΔΕΒΕ. Εμείς ε, είμαστε γνωμοδοτούσα Επιτροπή. Ο κ. Ταρό αντικαθιστά τον κ. Σολέ. Κύριε Ταρόν, είστε έτοιμος. Εξ ονόματος του συναδέλφου Τζόρντι Σολέ, που δεν είναι στη φυλακή, έχει, είναι απλώς άρρωστος, ε, θα σας παρουσιάσω τα πέντε σημεία τα οποία μου ζήτησε να αναφέρω. Η αναπτυξιακή η πολιτική πολιτική συνεργασία είναι βασικοί πυλώνε τη ε, υπηρεσία εξωτερικών εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση και την ευελιξία του τομέα 4, δεδομένου ότι τα πρόσφατα γεγονότα ε, δείχνουν ότι είναι περιορισμένε οι δυνατότητέ μα. Ε, το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία και το ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ σημαντικά για την ε, καταπολέμηση της κλιματικής ε, αλλαγής και για άλλους λόγους και έχουν συνεισφέρει να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικός παράγων αλληλεγγύης. Ο πρόεδρος σταματάει να μιλτεί και του ζητάει, του ζητάει να επιβραδύνει διότι μιλάει εξαιρετικά γρήγορα. Το σημειώνω λέει ο μιλτής, ε, η, εξωτερική, ανάθεση σε άλλες χώρες ε, της διαχείρισης των προσφυγικών ροών δεν είναι λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση που θα ακολουθείται από την υιοθέτηση συγκεκριμένων ε, δημοσιονομικών εργαλείων και επαρκών πόρων για να λυθεί η προσφυγική κρίση. Τέταρτο. Οι χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνία του Μπουζάν ε, θα είναι υπεύθυνε για την βελτίωση της ανάπτυξης, των πολιτικών ανάπτυξης και συνεργασίας και προσβλέπουμε σε περισσότερη συνεργασία. Η διεθνή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχύσει, να βελτιώσει την, ε, την καταπολέμηση της φτώχειας, ε, του αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Η τοπική και ανάπτυξη η, ε, και η ανθρωπιστική βοήθεια ε, είναι ε, στόχοι μιας βιώσιμης ατζέντα. Θα πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς προκειμένου να διαπιστώνουμε αν έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ. Καλή ανάρρωση λοιπόν παρακαλούμε να... Ε, καλή ανάρρωση στον κύριο Σολέ, παρακαλούμε να του μεταφέρετε τις ευχές μας και δίνω το λόγο στην κυρία Σουλίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον κύριο Τάραν, το οποίο τον εκπροσωπεί. Η πρόταση η Σολέ είναι μια καλή πρόταση. υπογραμμίζει τους βασικούς τομείς της αναπτυξιακής βοήθειας. Χρειάζεται να επενδύσουμε εδώ για να εκριζώσουμε την φτώχεια και να διασφαλίσουμε τη σωστή ανάπτυξη όλων αυτών των τομέων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ζωή των πολιτών, κάτι το οποίο θα βελτιώσει και την σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Να πω επίσης ότι η βελτίωση του κράτους δικαίου και της σωστής διαχείρισης είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και η δημόσια χρηματοδότηση φυσικά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα παράλληλα και τη σύνδεση ανάμεσα στην αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για να διασφαλίσουν την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά. Λοιπόν, θέλει κάποιος άλλος το λόγο κυρία Γουάρδια Ζάμπαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς στη Σοσιαλιστική Ομάδα συμφωνούμε 100% με την πρόταση την οποία κατέθεσε ο κύριος Σολέ. Νομίζω ότι περιγράφει με πάρα πολύ σωστό τρόπο τα μέσα συνεργασίας και αυτό είναι χρήσιμο και για την προετοιμασία του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου απαιτείται να υπάρξει μεγαλύτερη ε, συνοχή και διαφάνεια. Να διασφαλίσουμε λοιπόν περισσότερη διαφάνεια και συνοχή για τις πολιτικές ανάπτυξης. Ένα άλλο σημείο το οποίο έχει σχέση με την ευελιξία και τη χρηματοδότηση Μέσω αυτών των ταμείων προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές, να αντιμετωπίσουμε κρίσεις και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε ένα κάποιο περιθώριο προσαρμοστικότητας και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, ιδιαίτερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. βασικός στόχος αυτών των δύο μέσων είναι η συνεργασία ανάμεσα στην ανάπτυξη από τη μία και την ανθρωπιστική βοήθεια από την άλλη. Την αηφόρο ανάπτυξη. Για τη διαχείριση λοιπόν, όχι για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όχι για τη διαχείριση πολιτικών ασφαλείας, ούτε για τη διαχείριση της φύλαξης των συνόρων. Νομίζω ότι τα χρήματα αυτά πρέπει αποκλειστικά να πάνε προς την αναπτυξιακή βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γιούλαγκα, ευχαριστώ σύντομος θα είμαι. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την υποστήριξή μου στην πρόταση του κυρίου Σολέ, να υπογραμμίσω την ποιότητα της εργασίας του κυρίου Σολέ. Θα συμφωνήσουμε με τον συνδυασμό αυτών των μέσων και των ταμείων και τη συμπερίληψή τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε αυτές τις δύο πολιτικές και θα μπορέσουμε να καταστήσουμε πιο ευέλικτο το δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι ώστε τα ταμεία αυτά ούτε να μειωθούν ούτε να φυγούν με οποιοδήποτε τρόπο στο μέλλον. Να πω ότι συμφωνούμε επίσης και με τις ανησυχίες οι οποίες είχαν εκφραστεί και σε προηγούμενες εκθέσεις για τη συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανάμειξη αυτής της πολιτικής με τις συνοριακές πολιτικές και την πολιτική μεταναστευτική. Νομίζω ότι η ανάμιξη αυτή είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει σύγχυση και θα βλάψει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη τα μέσα αυτά να έχουν συγκεκριμένους στόχους στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών όπως τη Συμφωνία των Παρισίων για την αηφόρα ανάπτυξη, ε, για την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων και σεβόμενοι φυσικά πάντα στα πλαίσια της εφαρμογής τους την μεγαλύτερη, την υψηλότερη δυνατή συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Να υπογραμμίσω και εγώ την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε ο κύριος Σολέ και την εξαιρετική παρουσίαση του κυρίου Τάραντ. Άκουσα και τους συναδέλφους που ακολούθησαν και θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι όταν μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική και αναφέρομαι εδώ στα της Αφρικής, στην ουσία δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στο να στεγνώσουν ουσιαστικά οι πηγές από τις οποίες δημιουργείται η μετανάστευση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να τα αποσυνδέσουμε αυτά. Ο αφρικανικός πληθυσμός τα επόμενα 35 χρόνια θα διπλασιαστεί ένα δις 200 εκατομμύρια επιπλέον μικρών Αφρικανών. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα δεν μπορεί να, μας, να μη μας κάνει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν στον τομέα της μετανάστευσης. Κατανοώ αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σιουλάγα και η κυρία Γουαριαζάβαλ, αλλά όταν εγώ πάω στην εκλογική μου περιφέρεια και καταθέτω και εκθέτω μάλλον τις επιλογές τις οποίες έχουμε, νομίζω ότι στα πλαίσια της συζήτησης αυτής βρισκόμαστε ε, με υπεύθυνο τρόπο εν μέσω μιας πολιτικής η οποία έχει σαν στόχο να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές, δίδοντας τους Αφρικανούς την δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς στις χώρες τους και όχι να έρθουν εδώ. Αυτή είναι η μόνη παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω χωρίς να θέλω να ξαναρχίσει η συζήτηση. Λοιπόν, σταματήσαμε με τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Κύριε Τάραντ, θα θέλατε πάλι να πάρετε το λόγο εξ ονόματος του κυρίου Σόλε. Όχι. Θα σταματήσουμε εδώ. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 10 ε, το πρωί στις 20 Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 10 Μαρτίου και η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή Ανάπτυξης θα γίνει στις 20 Μαρτίου και στην Ολομέλεια του μηνός Απριλίου θα ψηφίσουμε ε, αφού συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βάιντερε. για τα πρωτόκολλα τα σχετικά με την αλληλεία και τις ε, οικονομικές εισφορές τις οποίες θα πρέπει να προβλέψουμε. Κυρία Βάιντερε έχετε το λόγο. Στο πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες ε, προφορτρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρώσει ε, συμφωνίες με πέντε χώρες στο στον Ινδικό Ωκεανό, Μαυρίτιο, Μοζαμβίκη, Μαδαρασκάρη μεταξύ άλλων και οι συμφωνίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί ή θα γίνουν διαπραγματεύσεις για αυτές. Έχουμε μία σύμπραση από το 1998 με το Μαυρίκιο ε, και φτάνουμε στην 30η ε, επέτειο ε, αυτής της ε, συμφωνίας ε, μας δίνει τη, τη δυνατότητα στο στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιάσει τόνο στην περιοχή και σε αντάλλαγμα η Ευρωπαϊκή, η, ο Μαυρίτιος, παίρνει χρηματικές αντιπαροχές για αυτό. Η περίοδος της, εφαρμογής του πρώτου πρωτοκόλλου έληξε στις 27 Ιανουαρίου πέρσι και ένα νέο υπογράφθηκε στις 26 Απριλίου πέρσι και θα ξεκινήσει ύστερα από την ολοκλήρωση της υιοθέτηση ε, και από τις δύο πλευρές. Αυτή η συμφωνία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, δεν αποτελεί μονόδρομο. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ε, έχουν γίνει σκέψεις από, το, από τις μεταρρυθμίσεις του 2013 σχετικά με την κοινή αλληλευτική πολιτική της διμερής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης των ε, κρατών έχουν αλλάξει το ε, μελλοντικό μας όρομα σχετικά με τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον περιλαμβάνει ε, ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο κοινό μας όφελος. Η επέκταση της συμφωνίας βασίζεται στις πρόστασεις της Επιτροπής Διαχείρισης τη Αλληλείας των του Ινδικού Ωκεανού και βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης ε, της προηγούμενης ε, συμφωνίας. Ε, μισό εκατομμύριο χρηματικής βοήθειας από το προηγούμενο πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκαν σε δράσεις για την βελτίωση της, του τομέα αλληλείας. Το νέο πρωτόκολλο 2017-21 θα, θα θα προσφέρει οικονομικές βοήθειες ε, ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, ε, δύο ε, 220.000 ευρώ προβλέπονται ε, για την υποστήριξη της αλληλείας ε, καθώς επίσης ε, και για την ανάπτυξη της οκεάνιας οικονομίας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά προβλέπονται οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη της οκεάνιας οικονομίας στον Μαυρίκιο Επίσης ε, θα ε, συνεισφέρει στην οικονομική του ανάπτυξη και κατά συνέπεια η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυρικίου ε, θα συμβάλλει την θαλάσσια οικονομία οι ε, χώρε που υποφελήθηκαν ιδιαίτερω ήταν η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίοι αποστέλουν λιευτικού στόλου ε, στον Ινδικό ωκεανό και θα πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε ότι η όρεξή μα για τον τόνο δεν θα εξαφανίσει τα αποθέματα τόνου ε, στι θάλασσε του Μαυρικίου. Θα πρέπει επίση να υπάρξουν οικονομικά εφέλη για τον εταίρο μα επικεντρωνόμενοι σε βιώσιμε πρακτικέ αλληλεία και από τη στιγμή που θα, θα ε, ολοκληρωθεί η συμφωνία με το Μαυρίκιο, θα ξεκινήσει ένα νέο πρωτόκολλο ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτηση και από τις δύο πλευρές. Ε, γι' αυτό το λόγο αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να σας καλέσω να υποστηρίξετε ώστε να δώσουμε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, σαφέστατα τα όσα μα είπατε. Δεν ξέρω αν κάποιο θέλει το λόγο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος. Ο κύριος Στάρεντ. Ε, θυμήθηκα το εξή ακούγοντας την συγκεντρία. Όταν ήμουν το 2000 στο Μαυρίκιο, ο υπουργό μου έδειξε μου έκανε μια ξενάγηση στον αλευτικό κλάδο και μου είχε πει ότι οι Σοβιετικοί ήταν αυτοί που είχαν ε, ζητήσει να αναπτυχθεί ο τομέα και η αγορά τους είχε καταρρεύσει. Ε, οπότε περίμενε και τη μόνη του ελπίδα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι φαίνεται είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Euh, Ιστορικό στοιχείο αυτό, ναι. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητά το λόγο. Για όσους αγαπούν τον να τρώνε τόνο, η συμφωνία είναι πολυθετική. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 26 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι. Όμως αυτές οι τροπολογίες δεν μπορούν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο. Η μόνη τροπολογία που μόνες τροπολογίες που μπορούν να γίνουν δεκτές είναι τροπολογίες απόρριψης του συνόλου του κειμένου. Η εισηγήτρια όμως μας ζητά να μην υποβάλουμε τέτοιου είδους τροπολογίες και συνεπώς να εγκρίνουμε τη συμφωνία. Οι μόνες αποδεκτές, παραδεκτές μάλλον, ε, τροπολογίες θα ήταν τροπολογίες απορρίψης. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα ψηφίσει ή 21-22 Φεβρουαρίου για το θέμα αυτό. Περνάμε στο επόμενο ζήτημα Ποιος άλλη είναι εδώ, οπότε θα μας παρουσιάσει την έκθεση του κυρίου Πάετ. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στη Μαγκοσμιοποίηση, αίτηση από τη Σουηδία Έριξον. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chair. Uh, I was Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριο Πρόεδρε. μου ζήτησε ο κύριος Παέτ να τον αντικαταστήσω. Η ε, Σουηδία ε, υπέβαλε μια αίτηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από τι απολύσει στην Έριξον. Ανέρχεται στα 210.000 ευρώ. Η υποστήριξη που ζητά είναι σημαντικό λοιπόν. Είναι η δεύτερη αίτηση της ε, Σουηδίας όσον αφορά της έριξον ε, υπήρξε μια αίτηση το Μάρτιο του 2016 ε, οι απολύσεις οφείλονται στην αρνητική ανάπτυξη ε, της ε, επιχειρηματικότητα στο hardware, καθώς επίσης και την αυξανόμενο ανταγωνισμό, ιδιαίτερω από την Ασία υπάρχει μία ασυμφωνία ικανοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων τη Ericsson και τη ζήτηση τη αγοράς και γι' αυτό το λόγο απολύθηκαν εργαζόμενοι. Και τέλος, πάνω από το 30% των ανθρώπων που απολύονται είναι στην ηλικιακή ομάδα 50 με 60 έχοντας ικανότητες που αφορούν συγκεκριμένα την βιομηχανία τηλεπικοινωνίας και γι' αυτό το λόγο κινδυνεύουν με μακροχρόνια ανεργία δεδομένης αυτή της αίτηση. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε άνθρωπους ε, οι οποίοι απολύονται από την Έριξον και να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν στην αγορά εργασία. Ο κ. Φερνάνδης ζητά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματο της Ιβάνα Μάλετιτ, που είναι απούσα, για να στηρίξω το αίτημα κινητοποίηση. για το ποσό των 2,1 εκατομμύριων ευρώ, 60% του συνολικού ποσού, για τα 900 άτομα που έχασαν τη δουλειά τους και ως συνήθως υποστηρίζουμε την χορήγηση βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους σε ένα καινούριο μια καινούργια θέση εργασίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ποιος άλλος θέλει το λόγο? Κανείς. Ωραία. Κύριε Άλλη. δεν έχετε κάτι να πείτε. μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, 6 ώρα το απόγευμα, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 21-22 Φεβρουαρίου. Δεύτερη έκθεση που αφορά κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτή τη φορά αφορά την Γαλλικία είδη ένδυσης. ο Γκοζάλης Πόντς θα έπαιρνε το λόγο, αλλά νομίζω ότι εκπροσωπείται από τον κύριο Μιλάν Μόν. Εξ ονόματος του συναδέλφου Γκονθάλεφ Πόντς θα σας παρουσιάσω την έκθεσή του. Πρόκειται για αίτημα κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για απολύσει τομέα της ένδυσης στην Ισπανία. Η Ισπανία επέβαλε έτοιμα για την κινητοποίηση του Ταμείου για να βοηθηθούν 303 εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους, ε, την εργασία τους από τον ε, Ιούλιο 16 στον τον Απρίλιο 17. Η Κομισιόν στις 6 Δεκεμβρίου 2017 ολοκλήρωσε την εξέταση και ε, απεφάνθη ότι καλύπτονται, ικανοποιούνται οι όροι. Η πρόταση αφορά 720.000 ευρώ, δηλαδή το 60% του συνολικού κόστους των δράσεων που προτείνονται. Αυτό το ποσό θα επιτρέψει στο σύνολο των απολυόμενων ε, να ε, δεχθούν την εφαρμογή μέτρων για την επανοδότηση της αγορά το γενεσιουργός αιτία των απολύσεων είναι η αυξήση των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την υπογραφή της, συμφωνίας, της Πολυελληνικής Συμφωνίας του 2004. Αυτό οδήγησε σε μείωση των τιμών και μια τάση μετακίνησης των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαλλική αυτό μεταφράστηκε σε σημαντική μείωση των επιχειρήσεων του υφαντουργικού κλάδου, 26% εξαφανίστηκαν από το 2010 έως το 2016. Πέντε επιχειρήσεις επηρεάζονται και οι πέντε στην επαρχία της Ακορούνια, στη Γαλλικία. Πρόκειται για μια ε, ε ζώνη της υπαίθρου, συγγνώμη, ε, που, της οποίας η ατμομηχανή, η βιομηχανική ατμομηχανή είναι αυτές οι επιχειρήσεις. Από το Δεκέμβριο 2016 ως τον Απρίλιο 2017 ε, η ε, παραγωγή μειώθηκε κατά 40%. Πρόκειται για άτομα περιορισμένων χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου και ηλικιών σχετικά μεγάλων. 303 άτομα, από αυτά 85,3% είναι γυναίκας, ηλικίας περίπου 30 με 54 ετών, κατά μέσο όρο. Η Ισπανία έχει προβλέπει έξι μέτρα, ε, Παρηματικό προσανατολισμό, ε, ε, αν αναζήτηση εργασίας κλπ. Έχουμε συντονιστεί με τις τοπικές αρχές και η αυτόνομη κυβέρνηση της Γαλλικίας θα είναι ο ενδιάμεσος οργανισμός διαχείρισης των ποσών. Τέλος, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις εκθέσεις, υπογραμμίζεται η σημασία ή το Ταμείο να μην υποκαθιστά τις επιχειρήσεις στις υποχρεώσεις τους ε, σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις και ε, υποχρεώσεις αναδιάρθρωσης. Η, η Ισπανία ικανοποιεί όλους τους όρους, συνεπώς ο εισηγητής μπορεί να θεωρηθεί, θε, ε, ε, ισχυρίζεται ότι μπορούμε να θεωρήσουμε πως είναι δυνατόν να υποστηριχθεί το αίτημα κινητοποίησης του Ταμείου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσω με προσοχή τις προτάσεις σας και θα τις μεταφέρω στον κύριο Γκονθάλεφ Πόντ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ συνάδελφοι. Ο Μπενίτο Ζιλουάγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω την κινητοποίηση του συγκεκριμένου ταμείου γιατί πράγματι επηρεάζει πάρα πολλούς ε, πολίτες, κυρίως γυναίκες στον τομέα ο οποίος μας ενδιαφέρει. Είναι σημαντικό λοιπόν να καλύψουμε την ανάγκη αυτή. Να κάνω τρία σχόλια. Το πρώτο αφορά το ίδιο το Ταμείο. Εμείς υποστηρίζουμε φυσικά την κινητοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του Ταμείου, όπως το έχουμε κάνει και στις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά θα ήθελα να επαναλάβουμε την κριτική την οποία ασκεί η ομάδα μας αυτής που λειτουργεί παρηγορητικά σχετικά σε σχέση με τις... Ε, por desgracia, en el sector de ε, empresas que son deslocalizadas para llevarlas a países. Εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να καλύψουμε την κατάσταση που δημιουργείται και η οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Ε, ξέρετε τι έγινε στο Μπαγκλαντές πριν δύο χρόνια με την κατάρρευση του κέντρου παραγωγής Πλάσα και θα πρέπει η ίδια η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολογηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το δεύτερο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι μιλάμε για το 83% ουσιαστικά των απολυμένων είναι γυναίκες. Η, ο τομέας της ένδυσης είναι ένας τομέας πραγματικά γυναικείος και υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους ε, μπορεί να υπάρξουν δυνατότητες κατάρτισης, ε, φροντίδας κοινωνικής, ε, διαχείριση των επιχειρήσεων επαγγελματικών, επίσης διαχείριση του ελεύθερου τομέα. Γενικά είναι τομείς στους οποίους η παρουσία των γυναικών είναι πάρα πολύ ισχυρή και μάλιστα ε, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προτείνονται ε, τέτοιου είδους μορφές κατάρτισης σε τομείς ε, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα, χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από την γυναικεία παρουσία. Τέλος νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε ένα τμήμα της βοήθειας αυτής να χρησιμοποιηθεί στην, συλλογικά στην εκπαίδευση και στη συλλογική εκπαίδευση των εργαζομένων αυτών. Η οικονομία στην παρούσα φάση στην Ισπανία Ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από ποσοστά επιδόσεων τα οποία είναι ε, καλύτερα από ό,τι σε άλλους τομείς και ταυτόχρονα οι συλλογικές μορφές επιχειρηματικότητας, ε, οι συνεταιριστικές δηλαδή μορφές αποδεικνύονται καλύτερες για τη διαχείριση τέτοιων ε, ε, δραστηριοτήτων όπως η επιπλοποιία είναι πολύ γνωστή η περίπτωση ανάληψης διαχείρισης ενός εργοστασίου επίπλων από ένα συνεταιριστικό σύνολο στην Βαρκελόνη. Νομίζω λοιπόν ότι η εκπαίδευση για συλλογικέ συνεταιριστικέ δράσεις είναι κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα θετικό για τον τομέα αυτό και είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν μια μορφή ενίσχυσης ενός τομέα ο οποίος δυστυχώ σε καθημερινή φάση μαστίζεται. και θα πρέπει φυσικά οι προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν να γίνουν συντονισμένα με ε, τους συνδικαλιστές και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της περιοχής. Θα ήθελε κάποιος να αντιδράσει στην έκθεση του Μίλαν Μόντς. Όχι. Είναι αλήθεια ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει μεγάλο βάρος. Αυτό το οποίο θα ήταν καλό είναι να προσαρμοστούμε στην παγκοσμιοποίηση για να αποφεύγουμε τις απολύσεις και όχι να περιμένουμε να γίνονται οι απολύσεις για να διαπιστώσουμε εκ των υστέρων ότι κάποιοι πολίτες έχουν χάσει πλέον την εργασία τους. Και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν από, τα, την ευρωπαϊκή επιδότηση γνωρίζουν ότι η Ευρώπη συμμετέχει στην διαδικασία επανακατάρτισής τους, γιατί περί αυτού πρόκειται τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά αναμειγνύοντάς τα με τις εθνικές δυνατότητες και τα εθνικά μέσα και συνεπώς δεν είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες συνειδητοποιούν πάντα την συμφωνία και την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς θα μείνουμε εδώ. Ο κύριος Μοντ δεν έχει κάποια συμπληρωματική παρουσίαση να κάνει. Εγώ θα μεταφέρω στον κύριο Γκονσάλες Πόν στις παρατηρήσεις σας Γνωρίζουμε τις οικονομικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, τις έχουμε συζητήσει και ξέρουμε επίσης ε, και τι έγινε με τη λήξη της συμφωνίας ε, ε, για, στον τομέα της ύφανσης γενικά και τι συνέπειες είχε όχι μόνο στην, Γαλλική, στην Γαλλική αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ε, οι πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται, οι διορθωτικές κινήσεις, ε, είναι συνδυασμός πολλαπλών μορφών και πηγών χρηματοδότησης και η βοήθεια για την, ε, για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες θα γίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Euh, Νομίζω ότι σε μια πρώτη φάση το ταμείο αυτό χρησιμοποιείται για τις απώλειες θέσεων απασχόλησης στον ε, βιομηχανικό τομέα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει και για τον εμπορικό τομέα σύντομα. Γίνονται κάποιες ε, αναδιαφρώσεις σήμερα. Ξέρετε ότι χάθηκαν 200.000 ε, θέσεις στον τομέα των μεγάλων σούπερ μάρκετ και κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή. Οι τροπολογίε θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 6η απογευματινή στις 5 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 21-22 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας. Ε, θα αναζητήσουμε τώρα τη συζήτηση για μία από τις συνέπειες του Brexit, δηλαδή την έδρα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής. Ο κ. Γκάιερ έχει το λόγο. αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κατά τη διαδικασία του Brexit θα πρέπει να σκεφτούμε σε την ε, μεταφορά των δύο ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βρίσκονταν στο Λονδίνο από τη μία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα αφορά τη μετακόμιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Γνωρίζετε ότι είναι μία από τις τρεις αρχές οι οποίες ασχολούνται με τα, με τα οικονομικά. Από την άλλη έχουμε την ΕΣ ΕΣΜΑ η οποία βρίσκεται στο Παρίσι και την Ιωιώπα που είναι στη Φραγκφούρτη ε, συμβαίνουν θαύματα. Πίστευα ότι το Συμβούλιο δεν θα κατόρθωνε ε, να ε, βάλει την ΕΜΠΑ σε μία από τις δύο βάσεις όπου υπάρχει ήδη μία παρεμφερής υπηρεσία αλλά ότι θα βρίσκαμε μία άλλη ενδιαφέρουσα πρωτεύουσα. Χαίρομαι όμως που είχα τελικά άδικο διότι τα καταφέραμε, το Συμβούλιο κατόρθωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να μεταφερθεί έρθει ε, στο Παρίσι. Ευτυχώς δεν έβαλα στοίχημα. Ε, τώρα όσον αφορά τα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ε, σημαντικό λοιπόν να τηρήσουμε ότι τα κόστη μετακόμισης ε, ε, θα, θα ε, ε, θα επιβαρύνουν τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το πώς θα διανεμηθούν τα κόστη του Brexit. Θυμόμαστε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της, του Ηνωμένου Βασιλείου είχε τη θέση ότι τίποτα θα ήταν το ιδανικό για μια συνεισφορά της Μεγάλης Βρετανίας προς τις υποχρεώσεις της ως όμως ένα κομμάτι της συμφωνίας είναι ότι τα κόστη της μεστακόμισης, ε, τα οποία είναι μεγαλύτερα για την ΕΜΑ από ότι την ΕΜΠΑ, ε, θα, θα ε, επιβαρύνουν τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ε, τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι αυτονόημο. Περιμένουμε λοιπόν από το νέο οικοδοσπότη από τη Γαλλία να βοηθήσει ούτω ώστε οι υπάλληλοι ε, να ε, διατηρήσουν τις συνθήκες εργασίας που έχουν ε, και κάτι ακόμα το οποίο θα συζητηθεί από τη συνάδελφο Χοτμάια είναι ότι αν αυτή αυτές οι δύο ε, υπηρεσίες που μοιάζουν ε, στις υποχρεώσεις τους βρίσκονται στην ίδια πόλη τότε προκύπτουν δυνατότητες συνεργίας. Θα μπορούσαν ίσως να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, το εκφράζω προσεκτικά, ε, θα μπορούσε να υπάρχει εξοικονόμηση στα τεχνολογικά, στην ασφάλεια, στην διαχείριση του προσωπικού. Όλα αυτά θα μπορούσαν να οργανωθούν από κοινού λοιπόν Οτιδήποτε λοιπόν πρακτικά δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο ε, της υπηρεσίας αυτή ε, και το τονίζω αυτό ε, θα μπορούσε να γίνεται από κοινού. Το τόνισα αυτό στην γνωμοδότηση και είπα ότι μπορούν να υπάρχουν πολλές συνεργίες σε περίπτωση που αυτό ήταν εφικτό. Θα πρέπει να το συγχρονίσουμε όμως ούτως ώστε οι δύο υπηρεσίες να βρίσκονται σε ένα κτίριο. Κάτι τέτοιο Όμω όμως δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Ε, μίλησα χθε με το διευθυντή της ΕΣΠΑ που ήδη βρίσκεται στο Παρίσι, το συζητήσαμε αυτό και μου είπε ότι δεν είναι τόσο εύκολο κάτι τέτοιο. Ε, τον έχουμε ε, να, να αναζητήσουμε νέα έδρα για δύο ε, υπηρεσίες. Η μία να μετακομίσει κάπου μέσα στο Παρίσι και μία θα έρθει από αλλού. Δεν είναι κάτι εύκολο. Βέβαια θα πρέπει ε, να ε, έχουμε υπόψη, μου, τον, υπόψη μας τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο Αυτό ε, αφορά, ε, αυτό λοιπόν τονίζω ιδιαίτερο στα όσα έχω ε, γράψει. Υπάρχουν όμως ανησυχίες και εδώ στο Κοινοβούλιο ότι μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να συμπτυχθούν αυτές οι δύο υπηρεσίες είναι μια ανησυχία που δεν συμμερίζομαι. Σε περίπτωση που γινόταν κάτι τέτοιο, αυτό θα γινόταν ύστερα από μια διαδικασία αξιολόγησης που θα πρέπει να συζητηθεί με την Κομισιόν για το αν θα έχει νόημα να γίνει όλο αυτό ε, και φυσικά υπάρχει και ο φόβος ε, ότι ε, μπορεί να συμπεριληφθούν και κομμάτια της υπηρεσίας στη Φραγκφούρτη. Όλο αυτό δεν συζητάται αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να έχουμε αυτή την φοβία. Το κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχει, όμως αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι αυτό σήμερα. Το θέμα αφορά να οργανώσουμε τη μετακόμιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και αν θα μπορούσε να γίνει επιτυχημένα και η Κομισιόν θα πρέπει να παρέμβει σε ορισμένες περιπτώσεις, να δώσει κατευθυντήριες, ε, να αναζητήσουμε από κοινού ε, για ακίνητα. Θα πρέπει τουλάχιστον να ε, προσπαθήσουμε ούτως ώστε όλο αυτό να γίνει πιο, όσο το δυνατόν πιο οικονομικά και χωρικά οι, υπηρεσία, οι υπηρεσίες αυτές να είναι κοντά. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν, ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε την Κομισιόν. Κύριε Σαλές. Ε, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού, Σαλές λέγομαι, πράγματι. Ε, συνεργαζόμαστε με τις άλλες δύο συναρμόδιες γενικέ διευθύνσει για να ε, παρακολουθήσουμε το θέμα από κοινού. Γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε το ότι θα πρέπει να γίνονται ε, εξοικονομήσεις κλίμακος μέσω συνεργειών προσπαθούμε αυτό να το παντρέψουμε με το κατάλληλο timing. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μετακομίσει το Μάρτιο 19, ενώ η ΕΣΜΑ λίγο πιο νωρίς. Οπότε υπάρχει μια διαφορά εκεί χρονική, αλλά προσπαθούμε να βρούμε μια μέση λύση. Πολύ δε περισσότερο που οι γαλλικές αρχές ε, μας ε, έχουν κάνει μια πολύ καλή προσφορά, ένα κτίριο ήδη και ε, διευκολύνσεις οικονομικές. Είμαστε σε επαφή με τις ε, δύο γενικές ε, διευθύνσεις στις οποίες αναφέρονται οι αρχές αυτές, οι υπηρεσίες αυτές και με τις Ολλανδικές και Γαλλικές αρχές αντίστοιχα. κυρία Βιώ έχει το λόγο. Euh, Άκουσα τα όσα μας παρουσιάστηκαν για τις σύνδικες εργασίας αυτών που θα εργαστούν στη Γαλλία. Θα ήθελα να ζητήσω μερικές διευκρινήσεις όμως δεν καταλαβαίνω πλήρως την παρατήρηση που αφορά το κόστος της μετακόμισης της αρχής. θεωρείτε ότι η Βρετανία θα πρέπει να λάβει ένα τμήμα του κόστου. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώ διαμήφθηκε από καλύτερα, τι ελέγχθη ακριβώ στι συζητήσει. Δεύτερον, τροπολογίε 3, 4 και 5 για τι συνέργειε. Ανάμεσα στην ΕΣΜΑ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το, η συζήτηση γίνεται σε τεχνικό επίπεδο, αν καταλαβαίνω καλά αλλά ίσως θα ήταν χρήσιμο να το δούμε και στην ουσία του πιο πολιτικά και να θέσω το εξή ερώτημα που πιστεύω ότι συνδέεται. Μας ικανοποιούν αυτή τη στιγμή οι κανονιστικοί μηχανισμοί για τις τράπεζες και το χρηματοοικονομικό τομέα. Ε, εγώ θα ήθελα να ενισχυθεί δυνατότητα ελέγχου των αγορών σύμφωνα με τη συζήτηση που κάναμε και σήμερα το πρωί για τον προπολογισμό. Πρόεδρος, η δεύτερη ερώτησή σας υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Κύριος Δοσάντος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με την πρώτη ερώτηση, das Σχετικά με τις, εξ, τις υπηρεσίες αυτές, τις εξωτερικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τις, ε, την ε, αρχή των τραπεζών, θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπατε βέβαια ότι ξεπερνά τις αρμοδιότητες της ε, Επιτροπής μας, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά το ερώτημα τίθεται να πω επίσης ότι έχω εμπιστοσύνη στον συνάδελφο Γκάιερ, ο οποίος έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, υπάρχουν πολιτικές ε, πλευρές, υπάρχουν τεχνικές πλευρές οι οποίες μεταξύ τους μερικές φορές είναι αλληλοσυνδυόμενες. Φυσικά είναι λογικό μια χώρα να ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση μιας τέτοιας ε, υπηρεσίας. Ξέρετε ότι είχαμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις στη χώρα μου για την αρχή ε, για τα φάρμακα. Η δημοκρατία έπαιξε τον ρόλο της και δεν επελέγει η χώρα μου επελεγεί Ολλανδία, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα πρέπει να δημιουργούν το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο και την ύψιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Πρέπει να γίνονται οικονομίες κλίμακας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα πρέπει και άλλα θέματα να ληφθούν υπόψη. Αυτό το οποίο πάντως έχει σημασία είναι ότι δεν θα πρέπει να γνωρούμε και τους εργαζομένους σε αυτές τις υπηρεσίες εγώ έχω εμπιστοσύνη στον εισηγητή, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια σωστή πρόταση. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να έχει ζητήσει το λόγο. Η κυρία Χόλμαϊερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. βρισκόμαστε εδώ για τα... Ε, δεν είμαστε υπεύθυνοι ε, για ζητήματα περιεχομένου, όμως είναι σημαντικό όσον αφορά τη συμμετοκόμιση ε, τη ΕΠΑ, δεν θα πρέπει ξαφνικά να έχουμε πάρα πολλά ζητήματα περιεχομένου, όπως είναι για παράδειγμα ποιε είναι οι λειτουργίες της κατάστοτε τράπεζες. Για μένα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει το αν θα βρίσκονται στο κοινό κτίριο ή σε διαφορετικά το σημαντικό σημαντικό είναι ε, να ε, είναι λειτουργικά και όχι να είναι ε, κτίρια πρεστίζ τα οποία θα είναι πανάκριβα και τα οποία θα, τα πληρώσει το Παρίσι επειδή τα θέλουν και καλά εκεί ή το αν θα βρίσκεται στις καινούργιες, στα καινούργια κράτη-μέλη. Δυστυχώς δεν μπορώ να αλλάξω την απόφαση που ελήφθη. Έχουμε περισσότερα ε, κράτη, ε, νέα κρατημέλη. Ο ασχέτως αυτού όμως ε, είναι σημαντικό όταν έχουμε να κάνουμε θέματα για κοινό προσωπικό, τότε θα μπορούσε αυτό και στις Βρυξέλλες να γίνει. Δεν χρειάζεται να θα μπορούσε να γίνει αυτό σε ένα κτίριο και θα πρέπει να προσέξουμε όμως τα κόστη και θα ήθελα να τονιστεί αυτό στο φάκελο. Ε, διότι ε, πάντα μας παρουσιάζονται τα πιο ακριβά πρότυπα και σίγουρα το Παρίσι μετά το Λανδίνο είναι ό,τι πιο ακριβό μπορούμε να φανταστούμε ε, και ύστερα από τις συζητήσεις που είχαμε τις υπηρεσίες με εξέπληξε το γεγονός ότι συνεχώς ε, είμαστε μόνοι ε, εγκαταλειμμένοι από την Κομισιόν όσον αφορά τις συζητήσεις ε, που κάνουμε με την Βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το τι βοηθάει και τι όχι και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να τονίσω η Κομισιόν να είναι συνυπεύθυνη ώστε να βοηθήσει τις υπηρεσίες τους διότι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν την ικανότητα μόνες τους να διαπραγματευτούν με την Βρετανική κυβέρνηση παρόλο που υπάρχει ο αντίστοιχος εταίρος για αυτό. νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα παίξει θα πρέπει να παίξει έναν ρόλο στις συζητήσεις με την Βρετανική κυβέρνηση. Πρόκειται ε, για ε, υπηρεσίες που έχουν τις δυνατότητες τους. Ε, ξέρω ότι έχουμε τη ΣΥΠΟΛ η οποία φεύγει από την Μεγάλη Βρετανία επειδή κατέληξαν στο ότι τελικά δεν τη θέλουν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, είμαστε περιορισμένοι όσον αφορά τις συζητήσει ε, με την ε, κυβέρνηση και ε, υπάρχει ανάγκη για βοήθεια και γι' αυτό το λόγο ζητάμε από την Κομισιόν να μην εγκαταλείψει αυτές τις υπηρεσίες. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα διότι δεν είναι δυνατόν υπηρεσίες όπως για παράδειγμα αυτή που εξετάζει τα φάρμακα ξαφνικά να πρέπει να κάνει διαπραγματεύσεις με την Βρετανική κυβέρνηση. Κύριε ε, Και εγώ έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Γκάιερ σχετικά με τα κόστη. Για να επιλέξουμε μία τοποθεσία θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθούν κάποια κριτήρια. Το κόστος λοιπόν ήταν ένα κριτήριο στην επιλογή της τοποθεσίας, ε, διότι άκουσα ότι και η Πορτογαλία για παράδειγμα ήταν μια πιθανή τοποθεσία. Σημερίζομαι τις ανησυχίες της Μόνικα ότι τα κόστη είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό το λόγο αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το Παρίσι, δεν είναι ιδιαίτερα φθηνό. Parce Υπήρχαν πολλοί υποψήφοι και οι διαπραγματεύσει κατέληξαν σε αυτόν, στο Παρίσι. Monsieur le rapporteur. Ο εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τι ερωτήσει, ε, Πράγματι, ε, δεν μπορώ να πω πολλά για τη διαδικασία διότι συζητήθηκε στο Συμβούλιο όλο αυτό. Και όταν λοιπόν το Συμβούλιο αποφασίζει για την έδρα ε, υπηρεσιών υπάρχουν κριτήρια τα οποία είναι αντικειμενικά ε, και ακολούθως υπάρχει και η πολιτική. Ε, και γίνεται μια ανάμειξη αυτών στο παρελθόν όσον αφορά ε, την, την έδρα. Είχαμε συζητήσει, έχουμε για παράδειγμα μια υπηρεσία που υπάρχει στην Κρήτη ε, και είναι δύσκολο κόσμος να πάει εκεί και επίσης δεν υπάρχει κανένα διεθνές σχολείο εκεί πέρα. Ε, η προσβασιμότητα και η δυνατότητα ε, για την εκπαίδευση όταν κάποιος ε, πάει με την οικογένειά του ε, σε μια νέα θέση εργασίας είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην όλη διαδικασία και βέβαια συνυπολογίζονται και τα κόστη. Είμαι σίγουρος ότι στη Γαλλία το ανέφερε η Μόνικα ότι σίγουρα μπορούμε να βρεθούμε πιο φθηνά ε, νίκια, ε, όμως ε, η εγκύτητα στην αγορά είναι ένα κριτήριο, η προσβασιμότητα ένα άλλο. Θα προτιμούσα και εγώ στην πατρίδα μου στην Έση ξαφνικά να δω μια υπηρεσία, όμως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα λάβουμε υπόψη μας όσον αφορά τα κόστη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το ερώτημα το κόστος ε, της ε, διαχείρισης και το ερώτημα σε, ποια, ε, σε ποιο ακίνητο θα βρίσκεται η υπηρεσία είναι ένα θέμα. Όταν έκανα μία από τις πρώτες μου επισκέψεις βρισκόμουν στη Βιέννη στο Schwarzenberg Ring το οποίο είναι μία αρκετά πλούσια περιοχή όταν περνάς ε, ως ε, Γερμανός ε, τουρίστας από εκεί και βλέπεις αυτό το παλιό παλάτι με την, ευρωπαϊκό, με την ευρωπαϊκή σημαία, η πρώτη αντίδραση είναι να που πάνε τα λεφτά μου λοιπόν. Ε, ένα μεγάλο κομμάτι του ενοικίου για παράδειγμα ε, καλύπτεται από την ε, Αυστρία και τη Βιέννη που το βλέπουν ως πολιτικοί να προσελκύουν διεθνείς υπηρεσίες στη Βιέννη. Πόσο ακριβό λοιπόν είναι εν τέλει το, το ενίκιο στο Παρίσι αφενός και αφετέρου το ανέφερε η Μόνικα ε, τι, ε, κατά πόσο θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης ε, από όλο αυτό. Ε, βέβαια όταν κοιτάζουμε τον ε, προϋπολογισμό ε, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ ακριβό. Το άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε αφορά την ανάληψη του κόστους από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί δεν γίνεται κάτι διότι ύστερα από την αποδοχή της πρώτης συμφωνίας σχετικά με, την, με τον Brexit η απόφαση ελήφθη. Πρακτικά λοιπόν γίνει ο λογαριασμός και ποιες υποχρεώσεις ε, θα έχει ε, η Βρετανία και ποιες όχι και συμφωνήσαμε λοιπόν ότι τα κόστη μετακόμισης των υπηρεσιών δεν θα βρίσκονται στις υποχρεώσεις της ε, Μεγάλης Βρετανίας, θα μπορούσαμε να το δούμε και διαφορετικά, όμως για άλλη μια φορά καθώς ακούμε βρετανικές φωνές εδώ μέσα που μας, ε, λέει, που μας λένε πόσο άσχημα η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, αντιμετωπίζει την, Ευρωπαϊκή, την Βρετανική κυβέρνηση και τον Βρετανό φορολογούμενο. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε στην, ε, στις εφημερίδες πώς θα ήταν για, μια για την άλλη υπηρεσία και ε, εκεί θα στην Ευρωπαϊκ... στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, πώς ε, θα γίνει η διανομή των κόστων εκεί πέρα. Ε, αυτά όσον αφορά τα ε, ερωτήματα περιεχομένου, αυτά δεν θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα, αλλά στην ΕΚΟ και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Πρόεδρος, η Κομισιόν έχει κάτι να προσθέσει? Όχι. Ναι. θέλουμε να κάνουμε κάποια σχόλια για τις τροπολογίες. Για την τροπολογία μόνο 1 περί των, του κόστους μετακόμισης που θα προτείνει να αναλυθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω θα πρέπει να διευκρινιστεί λίγο ακόμα το θέμα. Γιατί αυτό συζητείται αυτή τη στιγμή. Ε, μεταξύ της ε, ε, υπηρεσίας φαρμάκων και της Βρετανικής κυβέρνησης. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή των διαπραγματεύσεων, σας υπενθυμίζω, ήταν το κόστος να βαρύνει τις Βρετανικές αρχές. Αυτό μάλιστα είχε συμπεριληφθεί και στην προκαταρκτική συμφωνία της 8 Δεκεμβρίου. Οι Βρετανικές αρχές ε, δεσμευόντουσαν να διευκολύνουν τη μετακόμιση ε, συμπεριλαμβανομένης και της μείωση του κόστους. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Τροπολογία υπαριθμών 2. προτείνει να πάμε λίγο πιο μακριά από αυτό που προβλέπετε σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για τις έδρες των υπηρεσιών, μεταξύ ε, των υπηρεσιών και των εθνικών κυβερνήσεων. Καταλαβαίνουμε το στόχο, ε, κατάλληλες ε, συνθήκες και αποτελεσματικές λύσεις κλπ. Αλλά ο κανονισμός έτσι όπως έχει προταθεί νομίζω ότι καλύπτει τις συνήθεις πρακτικές σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες περί εδρών. Τέλος, για την τροπολογία 4 που αφορά το, την παράφο 3β της, ε, των αιτιολογικών σκέψεων που αναφέρεται ε, την ε, αυξημένη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και τις εργασίες της ε, διοργανικής ε, ομάδας για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοργανική ομάδα εξακολουθεί να συνέρχεται. Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι συστάσεις της, οπότε θεωρώ ότι η αναφορά σε αυτήν δεν είναι σωστή. Άρθρο 7, τροπολογία 5 τώρα, προτείνει να ενισχύσουμε τους στόχους ε, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. Αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από τις διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες. Δεν υπάρχει λόγος να υπογραμμίσουμε ξανά αυτό το στόχο στο διατακτικό του κειμένου νομίζω ότι προσθέτει κάτι στην ευκρίνεια του άρθρου. Πολύ δε περισσότερο που θα είναι, πιο δύσ... θα είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί η εφαρμογή του με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Έχετε κάποιες αντιδράσεις σε αυτές τις παρατηρήσεις. Καλώς θα σταματήσουμε τη συζήτηση αυτή εδώ. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 30 Ιανουαρίου 12 η ώρα. Περνάμε στην κυρία Χολμαϊερ γιατί θα συζητήσουμε πάλι για τις δύο αυτές αρχές. Μόνικα. Έχετε στη διάθεσή σας 13 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Έχουμε τρεις ε, συνολικά φακέλους ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συγγνώμη, ε, θα πάμε ε, στο έγγραφο εργασίας για την ΕΠΑ και την ΕΜΑ. Η ε, γαλλική κυβέρνηση λοιπόν μας έκανε μία προσφορά σχετικά με δύο κτίρια ε, είναι στο La και στο κέντρο της, ε, των Παρισίων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το La υπολογίζεται ε, στο Παρίσι, αν και δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά το λαμβάνουμε υπόψη μας, το ανέφερε και ο κύριος Γκάιερ. Η ΕΜΠΑ αναζητά κτίριο για ενοικίαση 12 χρόνων 4 με 5.000 ε, τετραγωνικών ε, εξετάζεται ε, να φιλοξενηθούν όλα τα, όλα, όλες οι υπηρεσίες στο Παρίσι σε ένα κτίριο, άρα δεν θα είναι μόνο το ΕΜΠΑ αλλά και το Ινστιτούτο Ερευνών Ασφάλειας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια έρευνα αγοράς. Το, Το αργότερο λοιπόν του Ιούνιο ε, του χρόνου θα πρέπει ε, να γίνει η συμφωνία για να ξεκινήσει αυτό. Θα είναι δύσκολο όλο αυτό. Ανυπομονώ να δω το τι μας περιμένει. Ε, επίσης θα ήθελα να πω ότι τα κόστη θα είναι ίδια με τα όσα ήδη υπάρχουν τα ε, έξοδα λοιπόν θα είναι ίδια ε, στο Λονδίνο και στο Παρίσι ε, και λαμβάνοντας υπόψη της προσφοράς της κυβέρνησης για 1,25 εκατομμύρια βοήθειας. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα είναι ετησίως και η κυβέρνηση θα πρέπει να τηρήσει τους κανόνες που θέτει υπομονώ να δω τι θα μας παρουσιάσουν λοιπόν όσον αφορά την, ε, τον οργανισμό φαρμάκων. Είναι ε, σημαντικό να υπάρξει ένα μεταβατικό κτίριο. Η ε, κυβέρνηση της Ολλανδίας λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να ε, ψηφιστεί όλο αυτό από το ε, Κοινοβούλιο και είπε η κυβέρνηση ότι θα ε, αναλάβει όλα τα κόστη διότι το αίτημά μας για μεταβατικό κτίριο ήταν ξεκάθαρο, είναι σημαντικό αυτό διότι στη συνέχεια το κτίριο Βιβάλτι θα πρέπει να δημιουργηθεί, να κτιστεί τα ε, στοιχεία, οι πληροφορίες ε, και οι ημερομηνίε θα μας δοθούν. Το κτίριο Βιβάλντι λοιπόν ε, θα ξέρουμε περισσότερα γι' αυτό από ότι και το Παρίσι. Θα έχει 28.500 τετραγωνικά μέτρα, θα υπάρχει ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο 400 τετραγωνικών μέτρων, ε, θα έχει 16 ορόφους ε, συνολικά ε, γνωρίζουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη εξωτερική κίνηση, πάρα πολλούς επισκέπτες δηλαδή, διότι ασχολείται με την πιστοποίηση των φαρμάκων. Έχουμε ένα πρόβλημα με το υπάρχον ε, κτίριο και χαιρετίζω την Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, για το γεγονός ότι ε, τότε είχαμε υποβάλει ένα πολύ αυστηρό working document το οποίο, το οποίο δηλώνει για ποιο λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του συμβολέου αυτό θα είναι αναγκαίο, θα ήταν αναγκαίο, ήταν μια παρανόηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονό ότι το Συμβούλιο, για το Συμβόλαιο ισχύει μέχρι το 39, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωση ε, διότι το Συμβούλιο είχε επιμείνει πάνω σε αυτό και δεν ήταν έτοιμο ε, να κάνει παραχωρήσεις και κάπου έπρεπε να πάει το αίμα και έτσι λοιπόν έπρεπε να το αποδεχτούμε. Το, η Επιτροπή μας είχε διαμαρτυρήσει διαμαρτυρηθεί για αυτό. Ή τα κόστη για την μετάβαση, για τη μετακόμιση λοιπόν είναι ξεκάθαρα ε, και ε, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε, ξαναλέω, αυτές τις δύο υπηρεσίες για να κάνουν τις διαπραγματεύσεις με τη Βρετανική κυβέρνηση καλό για άλλη μια φορά την Κομισιόν ε, να κάνει τις διαπραγματεύσεις μαζί με τις δύο υπηρεσίες ε, θα πρέπει να τονίσουμε και στην κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ότι εσείς θέλατε αυτές τις δύο υπηρεσίες τότε ε, και ε, τώρα αλλάξατε γνώμη, γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει να βοηθήσετε. Για το Κοινοβούλιο τώρα έχουμε, δηλώθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα ενός, η δυνατότητα υπενικίασης, κάτι το οποίο όμως, ε, μας, το οποίο όμως μας περιορίζει τις δυνατότητες που έχουμε λόγω του Brexit. Όμως ε, έχω, βρίσκεται σε μια πολύ καλή περιοχή, οπότε ίσως να βρούμε ε, έναν καλό υπενικιστή, αλλιώς ε, φοβάμαι για άλλη μια φορά όπως και επιβεβαιώθηκε ότι ε, θα υπάρχουν πολλά αυξημένα κόστη. Καλό την Κομισιόν επίσης να μας δώσει, να μας ενημερώσει ακριβώς ποια θα είναι τα κόστη και το, ποια είναι η στάση της, της Βρετανικής κυβέρνησης διότι όλο αυτό είναι αρκετά σημαντικό και γι' αυτό το λόγο έχω ζητήσει ένα έγγραφο εργασίας ε, ζήτησα, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ την γραμματεία μας ε, για τα έγγραφα τα οποία είναι πολύ καλά και θα μας βοηθήσουν ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ Τζέρμι. Όσον αφορά την ΕΜΠΑ λοιπόν θα ήθελα ε, να, ε, η δικαιοδοσία της ΕΜΠΑ και της ΕΣΠΑ να ε, διατηρηθούν και να μην δημιουργήσουμε μια υπηρεσία μαμούθ που θα έχει περισσότερες δικαιοδοσίες αλλά να υπάρχει διαφοροποίηση των υποχρεώσεων όπως αποφασίστηκε στο παρελθόν από το Κοινοβούλιο ε, το έγραψα ε, αυτό ε, ξεκάθαρα και ο Τζέρεμι είπε θα κρατήσει ακριβώς το πώς εξέφρασα ούτως ώστε οι συνάδελφοί της ΕΚΟΝ μου είπαν ότι το εκτιμούν. Είναι λίγο ασυνήθιστο αυτό σε ένα έγγραφο εργασίας όμως είναι ξεκάθαρο Επίσης όσον αφορά την κριτική ανάλυση των ε, δύο κτηρίων έχουμε ε, εγκρίνει ε, εμείς ως Επιτροπή αυτό και θα ήθελα να ζητήσω να παρακαλέσουμε την γαλλική κυβέρνηση ως νικητής του διαγωνισμού να διασφαλίσει ότι ε, θα υπάρχουν ε, λογικές συνθήκες συμφωνίες για τον νίκη και θα παρακαλούσα ε, τους συναδέλφους της Κομισιόν να μας ενημερώσουν εγκαίρως για τα κόστη και για τα επιπλέον κόστη που ίσως να προκύψουν. Επίσης η Γαλλία και η Ολλανδία θα υποστηρίξουν τις υπηρεσίες αυτές ε, κατά την μετάβασή τους ε, και ε, θα τηρήσουν τους, τους όρους τους οποίους παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή δάλλως της ο διαγωνισμός ήταν αυτός. το θέμα δεν αφορά μονάχα την γαλλική κυβέρνηση αλλά και την Ολλανδική κυβέρνηση. Έχει υπάρξει ένα ε, μικρό ε, λάθος ότι θα μπορέσουμε ε, να διασφαλίσουμε χαμηλά κόστη ενοικίασης. Αυτό δεν ισχύει μονάχα για τη Γαλλία αλλά και για την Ολλανδία. Θα ήταν μονομερές λοιπόν αν το αναφέρουμε αυτό, ε, καλούμε σε αυτό μονάχα την ε, γαλλική κυβέρνηση. Θα πρέπει, ε, έγινε λάθος λοιπόν, θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό και στην Ολλανδική κυβέρνηση. Επίσης όσον αφορά την αίμα και την συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές Ε, θα πρέπει ε, να βρούμε υπενικιαστή και ότι θα πρέπει να μείνουν τα κόστη χαμηλά. Η Κομισιόν παρακαλείται λοιπόν ε, να υποστηρίξει, βέβαια αυτό ισχύει και για την ΕΜΠΑ, και τα νέα σχέδια των κτίριων θα μας παρουσιαστούν εγκαίρως. Βρισκόμαστε σε μια ενδιαφέρουσα διαδικασία και θα υπάρχουν αρκετές συζητήσει πάνω σε αυτό. Η Κομισιόν το γνωρίζει αυτό, το γνωρίζουμε και εμείς αυτό. Euh, Ευχαριστούμε κυρία Συγγήτρια. Σοφές οι προτάσεις σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Κύριε Σαλές, από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ κρατάω τις συστάσεις της κυρίας Χολμάιερ ως ε, όργανο που προετοιμάζει τον προϋπολογισμό, τον επεξεργάζεται. Είναι σημαντικό να έχουμε σαφή εικόνα του πραγματικού κόστους των δύο μετακομίσεων. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή άλλωστε μαζί με τις υπηρεσίες και τις ε, δύο υπεύθυνε ε, αρμόδιες γενικές διευθύνσεις θα δοθούν διευκρινήσεις ε, και θα περιληφθούν στο τελικό έγγραφο που θα υποβάλουμε κάποια στιγμή το Μάρτιο ή τον Απρίλιο σε ό,τι αφορά τις μετακομίσεις για να βοηθήσουμε τις δύο αυτές αρχές τις συζητήσεις τους με τις εθνικές αρχές. <clears throat> λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι <clears throat> οι αρχές αυτές είναι αυτόνομες, ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Πρόεδρος, άλλες παρατηρήσεις, όχι, μπορούμε να... Α, και ο Στάραντ. Εν συντομία, πρόεδρε. Όπως πάντα συμφωνώ με τις συστάσεις για την πολιτική κτηρίων. Θα μπορούσε όμως η ισογήτρια να ελέγξει, να επιβεβαιώσει με την Κομισιόν το εξή. Αν στη Μόσχα έχουμε ένα κτίριο το οποίο, ε, το οποίο διοκτήτης είναι μια κυπριακή εταιρεία. Α, ακόμα είμαι στο Λονδίνο. Συγγνώμη, νόμιζα ότι τελειώναμε. Ε, εγώ πάντοτε είμαι πιο μπροστά από την εποχή μου. Ευχαριστώ κύριο Ταράν. Θα τελειώσουμε ακριβώς στις 5.30. για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Καταρχήν όμως σας κάνω μια δοκιμή των ηλεκτρονικών σας καρτών. Ε, άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Ah Donc nous avons 30, 30 euh, votants. 30 ψηφίσαντες, 30 οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, 31 με 30 ψήφους μόνο. Ένας από εσά έχει εισάγει κάρτα αλλά δεν έχει ψηφίσει. Θεωρώ όμως ότι η δοκιμή επέτυχε. La... Les premiers votes vont intervenir. Ψηφίζουμε καταρχήν την, ετήσια, την έκθεση Γκαρτία Θάβαλ σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκριση. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7, 8, 9 και 10. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11, 12 και 13 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επιβεβαιώνουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 17. Λήξη σουφορίας απορρίπτεται. 19 κατά 13 υπέρ. 17. Απορρίπτεται. Πάμε 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την 22 λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται 18 κατά 13 υπέρ 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Επιβεβαιώνουμε ηλεκτρονικά. Την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 17 κατά 15 υπέρ. Τροπολογία 26 κατά εποχές εγκρίνεται. Έκον παριθμών 12 καλύπτει από την 26. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές επιβεβαιώνουμε ηλεκτρονικά την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Για για... Ε, μία παραπάνω ψήφος για το ΕΛΚ. Ένας από εσάς παρακαλώ πολύ από το ΕΛΚ να αποσύρει την κάρτα του. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 12 κατά. είναι 28. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ε, επιβεβαιώνουμε όμως ηλεκτρονικά. 32. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 33. Εγκρίνεται 18 υπέρ 16 κατά. Έκον 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον όχι. Έκον 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Α, επαληθεύουμε. Λίγη. Εγκρίνεται. 18 υπέρ 16 κατά. Το τρι... Ήταν η 35 αυτή. έκονε 11 καλύπτει από 35. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 έχει αποσυρθεί. Έκον 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 καλύπτεται από την έκον 9. Τροπολογία 14, έκον 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39. Έχουμε προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 και 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 καλύπτεται, άρα καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 15, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προποφορική τροπολογία υπαριθμών 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έκον 25 καλύπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Έκον 22 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. εποχές Ας επαληθεύσουμε την 59. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Συγγνώμη, λέει 61 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι. Καταπίπτει. 62 καλύπτεται από την 63. 65 υπέρ κατά αποχές όχι καταπίπτει αυτή έκον 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67 με προφορική τροπολογία την υπαριθμό 4 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. απόχέ. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 18 υπέρ 16 κατά. 68 κατά πίπτη. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 73 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 72 υπέρ, όχι καταπίπτει. Έκον 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 74 δύο τμήματα. Θα χρειαστεί να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά εποχές καταπίπτει, απορρίπτεται. Το 75 υπέρ κατά αποχές ε, ας επαληθεύσουμε καλύτερα έναρξη της ψηφοφορίας λήξη 21 ψήφοι υπέρ, 13 κατά Εγκρίνεται, παρακαλώ πολύ να σηκώνετε πιο καλά τα χέρια σας. 76. Με προφορική τροπολογία την υπαριθμό 5 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 77. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Όχι, καταπίπτει αυτό το δεύτερο τμήμα. Το 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Επαληθεύουμε όμως. έναρξη Γιατί την 80. Λήξη. Εγκρίνεται. 18 υπέρ 16 κατά. 81. Υπέρ. Κατά. Λέω ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. λήξη της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Και πάλι επαληθεύουμε. Απορρίπτεται 17 κατά 16 υπέρ. Alors, dans ces conditions... Κάτω από τις συνθήκες αυτές θέτω το 82 σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ κατά. Αποχές δεν είναι ξεκάθαρο, θα ψηφίσουμε πάλι για την 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 18 υπέρ, 16 κατά. 87 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Ή ηλεκτρονικός έλεγχος για μια ακόμη φορά. Απερίφθη. 83. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ε, πολλοί δεν ψηφίζουν. Γι' αυτό λοιπόν για μια ακόμη φορά Ψηφίζουμε 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή 83. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 88 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Έκον 30. Έχει καταπέσει. 89 και 90 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 89 και την 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 18 υπέρ 16 κατά. 91 καταπίπτει. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή νομίζω. Όχι. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 93. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη 18 κατά 15 υπέρ. 94. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 96. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 95. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Επί της 95. Άρχεται. Πέρας. απερίφη, 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ψηφίζεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος πάλι. Τέλος. 19 υπέρ 15 κατά. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ο 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 100 με προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 101. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οι 103 και οι 104 έχουν, 104 έχουν καλυφθεί. 105 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκόν 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 107 υπέρ κατά, αποχές, απερίφη 108 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη 109 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 110 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 110. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 113 και 114 ταυτόσημες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά θα το ελέγξουμε. 113 και 114 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτές. Τροπολογία 116. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 118. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη 119 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 119 άρχεται πέρας απερίφθη 120 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 ρέτζι υπέρ κατά αποχές δεκτή 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή Έκον 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έκον 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Από την έκον 6, 7, 8, 21, 23 και 27 ομαδικά. Ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές δεκτές. Μετά έχουμε Ρέτζι 1, 2, 3, 4 και 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Το σύνολο του τροπολογημένου πλέον κειμένου ηλεκτρονική ψήφος. Τέλος. 30 υπέρ 3 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στον, στην εισηγήτριά μας. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Α, είναι σημαντική στιγμή για μένα και έχουν κατατεθεί κατατεθεί ορισμένε Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, απόχέ, δεκτή. 3 υπέρ, κατά, Αποχέ δεκτή. 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχή έχει καταπέσει η 8 γιατί έχει γίνει δεκτή η 9 10 υπέρ Συγγνώμη για μια στιγμή λέει ο πρόεδρο. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 11. Υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 14. Υπέρ. Έχει καταπέσει. Η 12 επίση Η 15 υπέρ.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 ηλεκτρονικός έλεγχος για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας, απερίφθη 19 κατά 15 υπέρ, 27 υπέρ κατά αποχές. Λοιπόν, απερίφθη για το σύνολο του τροπολογημένου κειμένου. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες 25 υπέρ 6 κατά 3 αποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ για την ε, προσπάθειά σας. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ε, έκθεση Esteban González Pons. Για την άμυνα. Οι 102, 124, 145 έχουν αποσυρθεί. Και οι 36 όπως και οι 61 τροπολογίες όλες αυτές απεσύρθησαν. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αν ψηφίζατε θα κερδίζαμε χρόνο περισσότερο. 78. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Μάλλον έχει καταπέσει 78. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 93 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 94 και 95 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθησαν. 96 υπέρ, κατά, έχει καταπέσει, μάλλον έχει καταπέσει. Θα ψηφίσουμε τώρα ομαδικά από την 96 μέχρι και την 100. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθησαν. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Η 102 έχει αποσυρθεί. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 104 υπέρ, Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 104. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απε, απερίφθη. 20 κατά 13 υπέρ. Αυτά για το 104. 105 και 107. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απερίφθησαν 106, 108, 169, 170 μαζί κατά αποχές απερίφθησαν συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική υπαριθμών 3 115 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 116 υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 116. Άρχεται. Πέρας. Απερίφη. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 137 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 138 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε για την 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Η 7 έχει αποσυρθεί. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 142 άρχεται. Πέραση τη Απερίφθη. 143. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απερίφθη. Συμβιβαστική 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Η 6 γίνεται δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εκατόν εξήντα Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ζητώ συγγνώμη. Ε, δεν είχα τον σωστό κατάλογο. Ζητώ συγγνώμη. 165. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 165. Ψηφίσατε όλοι οι της. Απερίφη. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 168 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115, 116, 117, 118 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται, απορρίπτονται. Ας επαληθεύσουμε όμως. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική παριθμών 10. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε αρχή της πιοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Παρακαλώ πολύ σηκώνετε καλά το χέρι σας να πάμε πιο γρήγορα. Και εγώ βέβαια που να προσέχω. Τροπολογία 28 καταπίπτει, 29 επίσης καταπίπτει. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 έχει αποσυρθεί 37 υπέρ καταπίπτει 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές Επαληθεύουμε λοιπόν. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. 40 υπέρ. Όχι το 40, η 40 Όχι. 40 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμό 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 46. 46 υπέρ. Όχι. Καταπίπτει γιατί έχει εγκριθεί ή έχει απορριφθεί 103. Και η 47. 48 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 49. Ε, καταπίπτει 50 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 51 Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 52. Καταπίπτει 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Καταπίπτει όχι. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική παριθμό 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 έχει αποσυρθεί 71 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 72 υπέρ έχει καταπέσει 73 επίσης συμβαστική υπαριθμό 18 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται ε, εγκρίνεται συγγνώμη το σύνολο του κειμένου τώρα Όπω τροποποιήθηκε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. 23 ψηφοί υπέρ, 10 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκονσάλε Πόνς. Ε, τμήμα 3 του προπολογισμού 2017 Υπάρχει αίτημα αναφοράς. Ε, Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι ε, η τελευταία μεταφορά ε, από τον ε, περσινό προϋπολογισμό και έτσι λοιπόν η υποχρέωσή μου ως γνωμοδότης δεν ε, είναι ε, ασύνηθε κάτι τέτοιο να μεταφέρονται τόσο πολλά ποσά, τόσο μεγάλο ποσά. Είναι θετικό παρόλα αυτά. Ε, υπάρχει κριτική για το γεγονό ότι δεν γίνεται χρήση των διορθωτικών προγραμμάτων. Εδώ έχουμε ποσά από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν μπορούμε να το ψηφίσουμε Υπάρχουν ε, επίσης μεταφορές ε, στην Frontex ε, καθότι η Frontex δεν έχει τη δυνατότητα τόσο γρήγορα όσο θα επιθυμούσαμε να προσλαμβάνει το προσωπικό της οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με όλα αυτό θα, θα ήταν ο παράγοντας συναλλάγματος ε, να μην γίνει ε, στο ε, ζλότι δεν συμφέρει κάτι τέτοιο είναι μεταφερές λοιπόν που είναι πολύ καλές και γι' αυτό το λόγο θα συνέστηνα στην Επιτροπή να ψηφίσει την συγκεκριμένη μεταφορά. Θέλετε να μας εξηγήστε λίγο αυτή την ε, τελευταία μεταφορά του χρόνου που είναι υψηλό ποσό, κύριε Ρέλ. Ε, αυτή η μεταφορά στο τέλος του χρόνου είναι μια δυνατότητα που δίνει το άρθρο 179 του Δημοσιονομικού Κανονισμού ε, στην Κομισιόν και επιτρέπει στην Κομισιόν να υποβάλει την Δημοσιονομική Αρχή μια πρόταση να μεταφέρει από όλους από όλα τα τμήματα του προπολογισμού της Κομισιόν ε, στα ε, προγράμματα ε, κοινή διαχείρισης για οποιοδήποτε ποσό πιστώσεων πληρωμών. Το ποσό για φέτος είναι 568 εκατομμύρια. Οι τρεις πιο σημαντικές πηγές αυτής της μεταφοράς είναι οι εξής. 50 εκατομμύρια στο Ταμείο για την Ευρωπαϊκή Βοήθεια για τους Απόρους. Ε, οι αιτήσει που είχαν έρθει από τα κράτη-μέλη ε, ήταν λιγότερες από όσες αναμέναμε. Δεύτερον, ποσό 86 εκατομμυρίων μπορεί να επιστραφεί από τον προϋπολογισμό του Ιουλίσα, της υπηρεσίας Ιουλίσα, εξαιτίας καθυστερήσεων στην υιοθέτηση νομικών βάσεων. Συνεπώς χρειάστηκαν λιγότερες πληρωμές κατά το 2017. Τρίτο μεγάλο κονδύλιο, 105 εκατομμύρια που δεν χρειάστηκαν στον προϋπολογισμό για το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική. Γιατί, γιατί στο τέλος περασμένου έτους απρόσμενα το ταμείο αυτό έλαβε σημαντικές συνεισφορές από τα κράτη-μέλη, συνεπώς δεν χρειάστηκε να κινητοποιήσουμε τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αρκετά υψηλές αυτές οι εισφορές από τα κράτη-μέλη ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του υπόλοιπου έτους. Πέραν, αυτού, έχουμε, πέραν αυτών έχουμε και αρκετά μικρότερα ποσά από 58 ε, γραμμές του προπολογισμού. Το συνολικό ποσό των 568 εκατομμυρίων ευρώ απορροφήθηκαν από το, απορροφήθηκε από το πρόγραμμα ανάπτυξη πέθρου γιατί η, τα αιτήματα ε, που ήρθαν από τα κράτη-μέλη για πληρωμές το τελευταίο τρίμηνο για την ανάπτυξη πέθρου ήταν πολύ πολύ ψηλότερες, ακόμα και από την πιο φιλόδοξη ε, πρόβλεψη της Κομισιόν. Αυτό, αυτό είναι πολύ καλά νέα πολύ καλή είδηση, διότι φαίνεται ότι τα προγράμματα εκεί πηγαίνουν πολύ καλά. Οπότε με αυτή τη μεταφορά, τέλος του χρόνου, μπορούν να πληρωθούν, να γίνουν αυτές οι πληρωμές ε, στη, χωρίς καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρατηρήσεις. Συζητά όλα ξεκάθαρα. Ωραία. Με ονομαστική ψηφοφορία Ψηφίζουμε. Λήξη ψηφοφορία. 24 ψήφι. υπέρ, μία κατά. Εγκρίνεται. Για το προορισμό του 2018 δεν έχουμε μεταφόρες. Για τα υπόλοιπα τμήματα, κύριε Σουάρτς, προϋπολογισμός 2018, κύριε Άσουαρτ, συγγνώμη, δύο τροποποιήσεις μας έχουν ζητηθεί πρώτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει να μεταφέρει 32 άτομα του προσωπικού μέσω της διαδικασίας Πασαρέλας για να γίνουν μόνιμοι. Είναι μια προσωρινή διευθέτηση για 9 μήνες μόνο. Είναι ε, ουδέτερο δημοσιονομικά, άρθρο 50 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τεχνικά, τυπικά δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, παρόλα αυτά εγώ συστήνω να εγκρίνουμε το ε, ε, συνέδριο ε, θέλει επίσης να μεταφέρει, μάλλον να ε, ε, να αλλάξει μία θέση AST8 σε AST-SE5. Ε, γιατί δυσκολεύονται να βρουν υποψήφιους για τη θέση AST8, γι' αυτό το λόγο θέλουν να τη μετατρέψουν σε SE5 στο Λουξεμβούργο. Δεν βλέπω καμία ανε... δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Και δύο μεταφορές και πάλι από το ελεκτικό συνέδριο θέλουν να μεταφέρουν 300.000 ευρώ από προσωρινό προσωπικό στην γραμμή άλλου, του άλλου προσωπικού εξωτερικές υπηρεσίες. Και πάλι είναι ουδέτερο δημοσιονομικά. Αυτό θα επέτρεπε όμως το Ελεκτικό Συνέδριο να ε, χρηματοδοτήσει ε, ε, την ασφάλεια των κτηρίων του και να αντικαταστήσει τρεις ε, υπαλλήλου ασφάλεια. Ο ένας είναι σε αναρωτική άδεια και πολύ καιρό και άλλοι δύο θέλουν, ε, είναι στι τεχνικέ υπηρεσίε. Είναι στι τεχνικέ υπηρεσίε και θέλουν να του μεταφέρουν. Ε, καλό αυτό διότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ασφάλεια στο συγκεκριμένο κτίριο. Ευχαριστώ, κύριε Ντεπρέ. Ε, δύο παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να μου εξηγήσουν, γιατί δεν κατάλαβα πολύ καλά, λέει ο κύριος Ντεπρέ εκτός μικροφώνου. Υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες θα μετατραπούν σε μόνιμες για την περίοδο που απαιτείται για το διορισμό των υπαλλήλων. Δεν καταλαβαίνω. Χωρίς μικρόφωνο ακούγονται κάποια σχόλια. Γιατί πρέπει να το κάνετε αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δεν γνωρίζω καλά τις διαδικασίες, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται κάτι τέτοιο. Είναι τεχνικό το θέμα. Σε εννέα μήνες θα επανέλθουν, εν πάση περιπτώσει, στην κανονική κατάσταση. Είναι τεχνικό το θέμα. Με φωτίσατε, λέει ο κ. Δεπρέ. Δεν ξέρω αν εκπρόσωποι της διοίκησης είναι εδώ, μπορούν να μας δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Εγώ ξέρω ότι οι συνεργάτες των πολιτικών ομάδων μπορούν ουσιαστικά να μονιμοποιηθούν ε, ε, ε, όταν γίνουν, όταν περάσουν στο κοινοβούλιο. Και στην ουσία απαιτείται για να επανέλθουν στις πολιτικές ομάδες η αλλαγή στο οργανόγραμμα. Αλλά υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου εδώ της διοίκησης. Κατάλαβα, λέει ο κ. Ντεπρέ. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων στα πλαίσια μιας διαδικασίας η οποία περιγράφεται εδώ πάρα πολύ συνοπτικά, οι οποίοι δεν μονιμοποιούνται, αλλά τελικά θα γίνουν υπάλληλοι, αυτό δεν μου λέτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λέει ο κύριος Ντεπρέ. Τι είναι αυτό του λέτε. Θέλουν να μονιμοποιηθούν, λέει ο πρόεδρος. Μα δεν υπάρχει κανείς που να εκπροσωπεί τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Ποιος είναι ο στόχος, να μπορέσουν να περάσουν στη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν όντας υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων, συνεργάτες των πολιτικών ομάδων και αυτή στιγμή μονιμοποιηθούν στο Κοινοβούλιο θα επανέλθουν στις πολιτικές ομάδες. Η μονιμοποίησή τους είναι ο στόχος, λέει ο Πρόεδρος, αλλά επιμένει ο κ. Ντεπρέ ποιος είναι ο στόχος. από τη Γενική Διάθυνση ΦΙΝ. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της διοίκησης του προσωπικού στόχος είναι πραγματικά οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων ή οι προσωρινοί υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων να μπορέσουν να περάσουν διαγωνισμό για να γίνουν υπάλληλοι. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουν ήδη μία θέση υπαλλήλου στην διοίκηση του Κοινοβουλίου και ή θα επανέλθουν στην πολιτική ομάδα ή θα περάσουν αφού περάσουν τον διαγωνισμό σε συγκεκριμένες θέσεις. Πρέπει λοιπόν για να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό να είναι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου και γι' αυτό έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό είναι ένα τμήμα της μεταφοράς. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε μονιμοποιούνται αυτοί που έχουν πετύχει στο διαγωνισμό και επιστρέφουν στις πολιτικές τους ομάδες μονιμοποιημένοι. Είναι μια τεχνική, αν θέλετε, ρύθμιση, η οποία είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος Ντεπρέ. Αν κατάλαβα καλά, η αρχική μου, αν θέλετε, εξήγηση ήταν σωστή. Όλες οι διαδικασίες αυτές γίνονται έτσι ώστε να μπορέσουν από την Πασρέλ να περάσουν στη δίκη του Κοινοβουλίου και να γίνουν μόνιμοι. Κοιτάξτε, πρέπει να, ε, χωρίς να είναι μέλη της διοίκησης του Κοινοβουλίου, δεν θα είχαν την δυνατότητα συμμετοχής. Οπότε γίνεται αυτή η τεχνητή, αν θέλετε, διαδικασία και καλό θα είναι η ε, διοίκηση του Κοινοβουλίου όταν παρουσιάζει τέτοια αιτήματα να δίνει περισσότερες εξηγήσει. Γιατί έτσι όπως είναι τώρα φαίνεται ότι γίνεται με σχετικά ελλειπτικό τρόπο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, ο μηχανισμός δεν ξέρω αν μπορείτε να τον εξηγήσετε. Να κάνω μια άλλη παρατήρηση, η οποία ίσως είναι και λίγο αστεία. Κοιτάξτε, ε, δεν θα έχουμε διευμηνία σε λίγη ώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ε, μπορεί να ζητήσουμε από τους διευμηνείς να μείνουν λίγα λεπτά παραπάνω. Να πω το εξής. Κοιτάξτε, είναι εδώ από τις δυόμιση οι διευμηνείς και έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, λέει ο πρόεδρος. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα, λέει ο κύριος Ντεπρέ. Οι διερμηνείς προσκαλούνται και στο κοκτέιλ που θα ακολουθήσει, ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε το λόγο κύριε Ερσέν. Θα είμαι σύντομος. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι προσωρινοί υπάλληλοι, οι οποίοι θέλουν να μονιμοποιηθούν. θέλουν να, περάσουν σε διαφορετικές μορφές μισθοδοσίας. Νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο η διαδικασία αυτή. Ε, εγώ δεν ήθελα να πω τίποτα τέτοιο. Εγώ απλά προσπάθησα να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Δεν πρόκειται εγώ να περάσω σε πολεμικές λαϊκίστικου τύπου. Euh, Κοιτάξτε, ο κύριος Σάσχουερθ ήταν σαφής. Πρόκειται για μια ρύθμιση την οποία θα μπορούσαμε να δεχθούμε έτσι κι αλλιώς και χωρίς να την ψηφίσουμε που λέει ο λόγος. Κύριος Σάσχουερθ. Κοιτάξτε, είναι κάτι πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε και να μην ψηφίσουμε. Στόχος ήταν να δημιουργηθούν οι θέσεις αυτές για το προσωπικό το οποίο είναι στις πολιτικές ομάδες και να μπορέσει να μονιμοποιηθεί στις πολιτικές ομάδες. Και μετά επιστρέφουν ακριβώς στις πολιτικές ομάδες, δεν παραμένουν στο κοινοβούλιο. θεωρητικά αυτοί εφόσον πετύχουν θα αποκτήσουν τη θέση της, τη μονιμοποίηση. Είπατε ότι είναι θέμα που αφορά το άρθρο 50, είναι κάτι το οποίο είναι ουδέτερο δημοσιονομικά, ως εκ τούτου προτείνω να γίνει δεκτή η πρόταση. Στην ουσία προτείνοντας να υπερψηφίσουμε, στην ουσία προτείνεται να μην ψηφίσουμε. Πολύ καλά. Ναι, λέει ο κ. Σάσχοθ. Καλώς λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας, αλλά αν θέλετε να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Η σύστασή μου είναι να εγκρίνουμε την πρόταση. Ναι, αλλά στα πρακτικά των συζητήσεών μας, αυτά τα οποία λέγονται εδώ θα καταγραφούν. Λοιπόν, πράγματι όλοι γίναμε σοφότεροι και συνεπώς η Επιτροπή Προπολογισμών εγκρίνει τις μεταφορές αυτές. Κυρία Χόλμαγερ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ε, τρία κτίρια αφορά τα ε, κόστη. Ε, βέβαια τα κτίρια αυτά έχουν νόημα. Έχουμε ένα κτίριο της, εξωτερικής Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, Δράσης. Η βελγική κυβέρνηση ζητά επιμήκυνση του, της ενοικίασης του κτίριου. έχει απορρίψει την ενοικίαση του κτίριου ΚΑΟ 15, οπότε θα πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό κτίριο το οποίο θα ενοικιαστεί μέχρι ότου να είναι διαθέσιμο το νέο νέο μεγάλο ε, κτίριο. Τα ε, κόστη συνολικά ε, θα είναι λίγο πιο ακριβά, όμως ε, καθότι θα έχουμε ένα υπάρχον κτίριο, τα συνολικά κόστη είναι στα 151 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ε, ενώ ε, στην Αυστρία είναι στα 166. Επίσης θα υπάρξουν ε, κόστη ανακαίνιση τα οποία πρέπει να γίνουν θα είναι το κόστος στα 500.000 ευρώ. Επίσης το, η ενοικίαση θα είναι στα τρία χρόνια. θα υπάρχει δυνατότητα επιμήκυνσης του ενοικίου. τα η έκταση είναι στα 5.000 τετραγωνικά μέτρα και θα ε, υπάρχει δυνατότητα ε, για το, θα υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας του ε, προσωπικού. Το δεύτερο κτίριο η ενοικίαση η παρούσα κατάσταση έχει ότι έχουμε τρία κτίρια γραφείων ε, στο Κόρτενμπεργκ. Η κατάσταση έχει ως εξής, ε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποχωρήσουμε ε, και χρειαζόμαστε καλύτερα κτίρια τα οποία Ε, θα ε, βρίσκονται σε καλύτερη, πιο σύγχρονη κατάσταση. Ε, έχουμε στα 6.700 τετραγωνικά μέτρα το, την υπηρεσία στρατιωτικής υποστήριξης. Έχουμε το CP στα 2.000 ε, τετραγωνικά μέτρα, το Crisis Management στα 1.700, το EPF στα 5.500 τετραγωνικά μέτρα, ε, το ε, Defense Building στα 5.000 ε, τετραγωνικά μέτρα και το IT, ασφάλεια IT στα 7.000 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε έχουμε μια υπηρεσία που αφορά την ασφάλεια. Όλα αυτά θα πρέπει να πάνε σε ένα νέο κτίριο. Ε, θα ε, πρέπει ε, να έχουμε ένα ειδικό συμβόλαιο το οποίο θα μας συμφέρει φορολογικά. Όλο αυτό θα κοστίζει λιγότερο. 21 χρόνια θα διαρκέσει. Η παράδοση του κτηρίου θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου του 2019. Όμως το συνολικό οι συνολικές αλλαγές και, με, ε, και ανακαινήσεις ε, θα ολοκληρωθούν ε, το 2020. Έχουμε μια έκθεση επίσης 18.000 τετραγωνικών μέτρων, έχουμε 550 εργαζόμενους. Το ενίκη ανέρχεται χωρίς έκπτωση ε, στα 4.500.000 ε, έχουμε επίσης ε, θα διαρκέσει για 21 μήνες μαζί με τη δυνατότητα μετάβασης θα μας δοθούν θα πρέπει να πληρώσουμε για 9 μήνες οπότε από το 2021 θα μπορούμε να το πληρώνουμε και η συνολική έκταση είναι στα 15.000 χρειάζονται επίσης θα πρότεινα λοιπόν να το ψηφίσουμε αυτό. Έχουμε ε, τα ζητήματα τα οποία αφορούν το κόστος της τεχνολογίας, το οποίο όμω δεν είναι ιδιαίτερα φθηνά, είναι απαραίτητα. Το νέο κτίριο συνολικά θα είναι πιο φθηνό από το παλιό κτίριο. 5 ε, εκατομμύρια... Ε, 25.000 ε, ε, και όσον αφορά ε, τις εκπτώσεις είμαστε πολύ καλά. Το νέο κτίριο λοιπόν καλύπτει όλα τα κριτήρια, κριτήρια ασφάλειας και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο θα πρότεινα να ψηφίσουμε υπέρ αυτού του σχεδίου. Αυτά τα δύο είναι συμπεριλάβουμε και τη Μόσχα που είναι διαφορετικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν, πάμε και στο κτίριο της Μόσχα. Ε, ο κύριος Τάου ενδιαφέρεται για αυτό ιδιαίτερος. Μέχρι στιγμής η κατάσταση ήταν ότι είχαμε ένα ε, όροφο που δεν χρησιμοποιούμε λόγω ε, ελάχιστου προσωπικού έπρεπε λοιπόν, θα το πω απλά, εξαιτία ε, το γεγονό ότι ε, θα ε, γκρεμιστεί το κτίριο, έπρεπε η πρεσβεία να αποχωρήσει και έτσι λοιπόν θα πρέπει να βγει από το κτίριο αυτό και να πάει σε, σε μια κανονική κατοικία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε για αυτό. Ε, με βάση την κατάσταση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η ε, κατάσταση λοιπόν έχει, έχει ως εξής, δεν μπορούμε να μένουμε σε ένα ξενοδοχείο, σε έναν ολόκληρο όροφο. Αυτό ε, μπορείτε να το φανταστείτε πως είναι για έναν Ευρωπαίο πρέσβη. έτσι λοιπόν μπορούμε να το ανακαινήσουμε, διότι ένα καινούριο κτίριο ως κατοικία θα είναι πάρα πολύ ακριβό και γι' αυτό το λόγο θα προσαρμόσουμε τον τελευταίο όροφο και θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε τόσο τον πρέσβη όσο και να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε τους απαραίτητους ε, χώρους ε, που χρειάζονται ε, όσον αφορά τις ε, συνθήκες ε, αποχώρησης έχουν αποφασιστεί και αυτές και τα κόστη αντιστοιχούν σε αυτό το οποίο θα περιμέναμε στην Μόσχα. Σας, θα ήθελα να σας πω ότι η κατάσταση για τον πρέσβη και για τους χώρους δεν είναι ό,τι καλύτερο και έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ένα χώρο που δεν θα ακούγεται από ε, οπουδήποτε αλλού. Και γι' αυτό το λόγο παρακαλώ να εγκριθεί όλο το νίκη ενέρχεται στα 2,392 εκατομμύρια ε, και ε, το συνολικό κόστος θα είναι 284. Θα σας καλώ να το ψηφίσουμε διότι και η ΑΦΕΤ μας ζήτησε να το επιταχύνουμε. Σας καλώ λοιπόν να το ψηφίσουμε. Τέσσερις θετικές νομοδοτήσεις λοιπόν. Κύριε Τάρεν, Ευχαριστώ ε, την εισηγήτρια, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι κατά ε, τι ιδέε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα πρέπει να έχει τι απαραίτητε τι εγκαταστάσει, αλλά όταν βλέπω το συμβόλαιο υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίε σχετικά με το ε, ποιοι είναι αυτοί ε, οι ε, Φέδων Γεωργιάδης και η κυρία Λαζαρίδου που είναι ε, υπήκοοι της ε, Κύπρου και είναι υπεύθυνοι για τα κτίρια στη Μόσχα, είναι η πραγματική Μήπω Μήπως θα πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ε, ιδιοκτήτε. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Θα πρότεινα, θα πρότεινα λοιπόν ε, να εξεταστεί το συγκεκριμένο θέμα. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον τον τελευταίο όροφο και δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο όσο έχει. θα διακοπεί από εδώ και πέρα η ελληνική διευμηνία. Καλησπέρα σας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 Oh, dis